ο κάποιο λάθος εδώ στις σημειώσεις μου. Ναι, όντως, είμαστε στο σημείο 8, που είναι η εξέταση των τροπολογιών όσον αφορά το πιστοποιητικό επιπλέον προστασίας για φαρμακευτικά προϊόντα. Ο εισηγητής, ο κύριος Λουίς Γκράντε Πασκουάλ, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής είχα την δυνατότητα να σας παρουσιάσω ως εισηγητής πώς ε, έβλεπα το πώς θα αντιμετωπίσουμε την έκθεση αυτή, η οποία αυτή καθ' αυτή έχει ένα μικρό βεληνικές, όμως είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ως προς το αποτέλεσμα που μπορούμε να πετύχουμε Το είχα πει και συνεχίζω να το πιστεύω ότι αυτό το θέμα που έφτασε αργά στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, δεν ε, ήταν ε, λόγω ή μη επιθυμία της Επιτροπής, αλλά ήταν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκό θέμα και αργήσαμε πολύ στο να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια εξισορροπημένη θέση και λογική από νομική σκοπιά. για να δίνεται η δυνατότητα στους ε, παρασκευαστές γενώσιμων και βιομηοδών να μπορούν να ανταγωνιστούν επιτυχώς με τις ε, τρίτες χώρες όταν λήξει η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Επίσης, είχα δηλώσει ότι υπάρχει ένα συνασπισμός από ό,τι φαίνεται μεταξύ δύο ομάδων κρατών που είναι περισσότερο υπέρ των γενοσύμων, γιατί εντό των κρατών αυτών έχουμε παραγωγή γενοσύμων και άλλων χωρών που είναι περισσότερο υπέρ των καινοτόμων φαρμάκων και Οι επιχειρήσεις αυτές ε, είναι κατεστημένες στη δική τους επικράτη, έχουν προβεί σε μεγάλες επενδύσεις και ουσιαστικά έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο για τα νέα δραστικά συστατικά που έχουν βελτιώσει την παγκόσμια υγεία. Επίση είχα πει και το περιλαμβάνω και στη συνέχεια θα αναφερθώ στι τροπολογίες ότι δεν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία ψευδή συζήτηση Δηλαδή να λέμε ότι τα γενώσιμα ουσιαστικά υπερασπίζουν και τους πιο αδύναμους και το να υπερασπίζουμε τους κοινοτόμους ε, σημαίνει ότι υπερασπίζουμε κάποιες θέσεις κυριαρχίας. Είναι παλιά η συζήτηση αυτή, η εξέλιξη των γενοσύμων ε, στον ε, παγκόσμια υγεία έχουν σημειώσει μείωση των τιμών, σημαντική πρόοδο και με αποτελεσματικό τρόπο έχουν φτάσει σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλές ομάδες και συλλογικότητες που στο παρελθόν δεν είχαν πρόσβαση στα φάρμακα. Η Παρασκευή των Γενοσύμων ε, σήμαινε μια παγκόσμια πρόοδο. Η πρόθεση της Κομισιόν με την τροποποίηση του κανονισμού ουσιαστικά θέλει να ευνοήσει τους παρασκευαστέ των γενοσύμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν επιτυχώ να ανταγωνιστούν και μίσες ευκαιρίε με τις ε, τρίτες χώρες που είναι απόλυτα, και να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι να ανταγωνιστούν τους παρασκευαστές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία κτλ. Προκύπτει ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ανατολικές χώρες που ε, ουσιαστικά επιδίδονται περισσότερο στην παραγωγή γενοσύμων και αυτό δεν είναι ένα δεδομένο που είναι υπέρ ή κατά, είναι ένα γεγονό και υπάρχει ένας συνασπισμός που μπορεί να μας διαιρέσει με ένα τρόπο ανεπιθύματο. Ε, δηλαδή, κάποιες ε, χώρες ε, να βρεθούν στο περιθώριο. Η πρόθεσή μου είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο συμβιβασμό όπου τα μεγάλα θέματα να έχουν οριστεί. Και εγώ στην έκθεσή μου έχω βάλει τα δυνατά μου έτσι ώστε να ευνοήσω πέρα από την προσπάθεια της Κομισιόν να ευνοήσει τους υπερσκευαστές των γενοσύμων αλλά χωρίς να απολωτριώσουμε τα νόμιμα δικαιώματα των παρασκευαστών καινοτόμων φαρμάκων που προφανώς έχουν κάνει τη δουλειά τους και έχουν δικαιώματα προστασίας ε, βάσει διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τώρα, εδώ, ερχόμαστε εδώ για να εξετάσουμε τις τροπολογίες που παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο. Είχαμε συνολικά 271 τροπολογίες, 22 ε, για τα εκτιμώντας και τα υπόλοιπα για το διατακτικό. Θέλω να αναφέρω ότι η προστασία του πιστοποιητικού δεν φέρει ε, καμία επίπτωση στην προστασία του συμπληρωματικού πιστοποιητικού ε, για τα προϊόντα παράγοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει αυτό. Δηλαδή οι κάτοχοι θα πρέπει να διατηρούν την αποκλειστικότητα και γι' αυτό η πρόταση συνοδεύεται από ασφαλιστικέ δικλείδε που εγγυώνται τη διαφάνεια και αποφεύγει ε, να υπάρχει παρέκκληση για την αγορά γενοσύμων και βιομοιδών. Ε, θέλουμε να έχουμε μια ισορροπημένη θέση εδώ. Υπάρχουν ε, τρία κυρία θέματα στην πρόταση και ελπίζω να μπορέσω να εργαστώ με όλους. Φυσικά θα ακούσω ε, τις διάφορες προτάσεις με πολύ προσοχή για να δούμε αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη θέση. Θέλω να πω εκ των προτέρων ότι η θέση της ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου είναι αρκετά κάθετες και δεν θέλουν να αλλάξουν την αναλογία αυτού του κανονισμού. Εγώ το κατανοώ αυτό και όπως θα δείτε στην εκθεσή μου έχω υποστηρίξει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ε, βέβαια, υπό την επιφύλαξη να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις που θα μπορέσουν να ευνοήσουν ε, τους παρασκευαστές γενοσύμων λίγο παραπάνω από αυτό που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω ότι σε τροπολογίες ε, υπάρχουν συμπτώσεις, ότι πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση ε, στον κάτοχο του ε, διπλώματος, γιατί εδώ μιλάμε για μια εξαίρεση σε δικαίωμα και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες και αληθινές πληροφορίες ε, προκειμένου να μπορούν να έχουν επαρκείς αποδείξεις για να παρουσιαστούν ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση. Ένα άλλο θέμα είναι η εφαρμοσιμότητα της πρότασης. Η διανοητική διοκτησία είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μία άμεση εφαρμογή του κανονισμού θα έπλητε δικαιώματα που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι. Γι' αυτό εμεί προτείνουμε εφαρμογή σε τρία-τέσσερα χρόνια ανάλογα με τη δημοσίευση του κανονισμού που εγγυάται την ε, σημασία να αντιμετωπίσετε το συντομότερο τα προβλήματα και από την άλλη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, θεσπίζοντας μια ομοιόμορφη ημερομηνία εφαρμογής και μια ε, μακρά μεταβατική περίοδο προκειμένου να εγγυώνται να εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων επενδύσεων. Έχουν δηλαδή ε, οι διάφοροι πρωταγωνιστές ε, έναν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν. Και βρισκόμαστε ε, όλοι τώρα στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αποθήκευσης, stockpiling. Stockpiling ε, σημαίνει ε, όχι μόνο αποθήκευση, αλλά πηγαίνει ακόμη πιο πέρα. Δηλαδή υπάρχει η πρόθεση να αναγνωριστεί η πρόταση της Κομισιόν. Γιατί ένα είναι να παρασκευάζει κανείς και να αποθηκεύει, έτσι ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικά με τις τρίτες χώρες και να μην ε, δίνει πλεονεκτήματα σε άλλους και άλλο είναι ε, κάτι που πηγαίνει πιο μακριά και είναι το νόμιμο συμφέρον. Θα πρέπει να δούμε ότι από την πρώτη μέρα υπάρχει δυνατότητα τα γενώσιμα να μπορούν να ανταγωνιστούν ε, στην εσωτερική αγορά της Ένωσης. Ε, αυτό είναι το κλειδί εδώ. Κανένας ε, δεν θέλει εδώ να εξαπατήσει και εγώ το λιγότερο. Έχω μιλήσει με όλους ε, και έχω ελέγξει ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Μίλησα με την Κομισιόν, με το Συμβούλιο, σε ποιο βαθμό θα ήταν δυνατόν κάποιο συμβιβασμός που να περιλαμβάνει κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες και να μην επιτρέπει να πετύχουν αυτό το στόχο που νόμιμα επιθυμούν οι παρασκευές γενοσύμων. Βέβαια βρίσκω μια φυσική δυσκολία. Είναι το προηγούμενο και φυσικό δίκαιο των ε, παρασκευαστών καινοτόμων φαρμάκων που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις. Σε αυτά τα πέντε χρόνια, αυτά τα πέντε χρόνια που τους δίνονται ε, για να εκμεταλλευτούν την επιτυχία του φαρμάκου, στην πρόταση της Κομισιόν, ε, ας το Τι κάνουμε με την πρόταση της Κομισιόν, τελικά ευνοούμε τα γενώσιμα. Έτσι ώστε ταυτόχρονα να μπορούν αυτοί οι παρασκευαστές να παρασκευάζουν γενώσιμα και να τα αποθηκεύσουν και να είναι έτοιμοι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Κοιτάξτε, έτσι είναι, αλλά είναι αδικία. Τα γενώσιμα να μπορούν να επιβληθούν. Τελικά ευνοούνται εδώ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα δεχτούν οι άλλοι παρασκευαστές των καινοτόμων φαρμάκων, ε, γιατί ουσιαστικά τους αφαιρείται ένα δικαίωμα που είχαν, ε, δηλαδή να εκμεταλλευτούν και να αποδώσουν επενδύσεις τους. Γιατί οι καινοτόμοι παρασκευαστές λένε δικαίως δεχόμαστε αυτό που θέλει η Κομισιόν. Μάλιστα ε, δεχόμαστε και τα όρια που θέτει η εκθέση του συγητή, αλλά δεν θέλουμε να πάμε πιο μακριά. Μας φαίνεται ότι είναι άδικο να πάμε πιο μακριά. Αν ε, φτάσουμε στα όρια θα πάμε σε αδιέξοδο. Όλοι ξέρουμε ότι το χρονικό πλαίσιο που έχουμε για να εργαστούμε είναι πολύ περιορισμένο. Ή θα βρούμε ένα συμβιβασμό που να είναι χρήσιμος. Ε, έτσι ώστε και το Κοινοβούλιο, δηλαδή και οι τρει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι Κομισιόν, να δεκτούν μία μορφή διεξόδου. Διαφορετικά, ε, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και θα ήταν αδύνατο να επιζήσει η πρόταση αυτή. Και αυτό είναι λυπηρό. Αλλά εγώ πρέπει ειλικρινά να το πω. Γιατί θα μιλήσω με όλους όσους κατάστατροπολογίες, με όλους τους ένα προς ένα, να δούμε ε, ουσιαστικά αν θα ε, κατέβουν στα χαροκόμματα, τέλο πάντων ε, θα επιμείνουν όσοι προβαίνουν σε Παρασκευή καινοτόμων φαρμάκων και να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε μακριά με τις ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το λέει και η Επιτροπή, μια μεγαλύτερη διάβρωση των δικαιωμάτων του πιστοποιητικού θα έστειλε ένα ενδικό μήνυμα σε άλλους εμπορικούς εταίρους με τους οποίους διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα δικαιωμάτων διανοητικής διοξίας. Δηλαδή εδώ επιστρέφουμε ε, στο θέμα της επεράσπισης ε, των αρχών που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, μία εξαίρεση της αποθήκευσης για να βελτιώσουμε την ταχύτητα θα πρέπει να είναι να, σε προ... λάμβει υπόψη και άλλου παράγοντε, όπως το μέγεθο τη αγορά, την ανταγωνιστικότητα τη αγορά, τι τιμέ, ε, τι αποζημιώσει. Αναφυσβήτητα τα στοιχεία αυτά έχουν σημαντικό ρόλο. Τελειώνω όταν ε, αναλύονται οι συνέπειε μια γενική κατάσταση, ε, δεν φαίνεται να είναι ο κύριο παράγοντα το πιστοποιητικό. Αλλά φαίνεται ότι οι τιμέ και αποζημιώσει είναι τα κύρια που καθορίζουν πότε το γενώσιμο μπορεί να μπει και σε ποια αγορά. Λαμβάνοντα υπόψη του συμβιβασμού, εγώ θα προσπαθήσω να συνομιλήσω με όλους, με όλους τους συντάκτες των ε, τροπολογιών και φυσικά ναι, θα χρησιμοποιήσω την καλή μου βούληση για την επίτευξη συμβιβασμού. Ένα συμβιβασμό που μπορεί να μπορέσει να αυξήσει την αντιγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Να βρούμε μία ισορροπία, να διατηρήσουμε ελκυστική την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, κέντρο ε, καινοτομίας ε, και καινοτόμων επενδύσεων και από την άλλη να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα των παρασκευαστών γενοσύμων και βιομοδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντα τι συνθήκε για να μπορούν να ανταγωνιστούν με ίσου κανόνε στι παγκόσμιε αγορέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι μάλιστα ο κοινό παρανομαστή όλων των συντακτών τροπολογιών που υπερασπίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα των γενοσύμων μετά από την Day One την πρώτη μέρα εισόδου. Εγώ νομίζω ότι είναι νόμιμα τα αιτήματά τους, όμως βλέπω ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο να γίνουν αποδεκτά από το άλλο μέρος και από την ίδια την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Φυσικά σέβομαι όλες ε, τις απόψεις και προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, ε, να μην είμαι υποπόλεως γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί κάθε αλλαγή που θα κάνουμε, ακόμα και στο μικρό κόμμα, έχει ε, επίπτωση σε πολύ μεγάλα συμφέροντα. Και βλέπετε ότι άλλε ευκαιρίε υπάρχουν σε άλλε χώρε, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να πούν: κάνουμε όλε αυτέ τι επενδύσει για να έχουμε ένα νόμιμο στόχο και έχουμε δικαίωμα να υπερασπίσουμε τι θέσει αυτέ. Αυτή είναι η θέση μου, κύριε Πρόεδρε, υπό την επιφύλαξη να αναλύσουμε μία-μία τι τροπολογίε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ δουλειά. Σήμερα κάνουμε μία γενική συζήτηση. Εγώ θα προβώ σε μεμονωμένες διαβουλεύσεις με τους συντάκτες των τροπολογιών και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε κάποιους συμβεσμούς, αφού όλοι θα έχουν αναλύσει το κατά πόσο είναι βιώσιμες οι προτάσεις τους. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λετόφσκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι τροπολογίες ε, οι οποίες κρατάθηκαν από το ECR έχουν ως σκοπό να επεκτείνουν το πεδίο της εφαρμογής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων στην προσβατησιμότητα σε σύγχρονα γενώσιμα φάρμακα, όχι μόνο σε πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός λοιπόν αυτών δεν, θα αφορά πλέον μόνο τις εξαγωγές στην Αφρική, αλλά θα καλύπτει και ανάγκες στην Ευρώπη που είναι τεράστιες. Τα φάρμακα με επιπλέον πιστοποίηση για εξαγωγή έχουν επιπλέον οικονομική αξία. Η πώληση στην εσωτερική αγορά έχει να κάνει με την ασφάλεια των ε, Ευρωπαίων ασθενών. Ελπίζουμε με τις διαπραγματεύσει να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι ευνοϊκή και για τους ε, ασθενείς αλλά και για τους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς τέτοιων φαρμακευτικών προϊόντων. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε στη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φόλκαμεν. Βέλκεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε, και θα μιλήσω γερμανικά. Σας ευχαριστώ για την ε, ενδελεχή ε, παρουσίαση. Και εγώ έχω σκοπό και ως πρόθεση να πετύχουμε μια γρήγορη συμφωνία. Ωστόσο, πιστεύω ότι αν το πετύχουμε αυτό στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αποτανθούμε και στην Ολομέλεια. Και αυτό θα θέλαμε να παραμείνει ως δυνατότητα, γιατί αυτά που άκουσα σε εξήγηση με σοκάρουν. Έχουμε ασχοληθεί από σε δύο επιτροπών με το θέμα αυτό και έχουμε δώσει το θέμα αυτό και στην Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για θέματα υγείας και ε, στην ψηφορία στην Επιτροπή αυτή ήταν συντριπτική η πλειοψηφία των συναδέλφων που υπερψήφισαν το συμβιβασμό. Ο συμβιβασμό αυτός λοιπόν πιστεύω ότι μάλλον η ευρεία συνένεση υπέρ του συμβιβασμού αποτυπώνει την επιθυμία του Κοινοβουλίου. Η παραγωγή γενώσιμων λοιπόν φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να πάρει ένα κίνητρο. Αυτό δεν το πετυχαίνουμε με την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να δώσουμε πλέον κίνητρα. Και εδώ βασικό θέμα είναι το stockpiling, η αποθήκευση. Χωρί το κομμάτι αυτό δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση για το συμβασμό της Επιτροπής. Ε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ το επιχείρημα των ε, ε, εμπορικών συμφωνιών που θα έβλεπτε το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα των ασθενών. Και τόσο σύντομα πριν από τι ευρωεκλογέ, θεωρώ ότι θα ήταν πραγματικά μοιραίο λάθο να αφήσουμε την ευκαιρία αυτή να φύγει από τα χέρια μα. Το θέμα του stockpiling λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει, θεωρώ, να. Αν χρειαστεί να ρωτήσουμε την ε, άποψη των συναδέλφων. Έχουμε λοιπόν τέσσερα σημεία τα οποία μας βρίσκουν, δεν μας βρίσκουν ε, σύμφωνο στο θέμα του stockpiling, το παιδί εφαρμογή ε, τη ε, ενημέρωση των παραγωγών όταν ξεκινάει η παραγωγή ενό φαρμάκου. Νομίζω ότι σε όλα αυτά τα θέματα θα μπορούσαμε να βρούμε μια ισορροπημένη λύση αν κάνουμε βήματα προς τα μπροστά και στο θέμα της ενημέρωση ε, είναι φυσικά πολύ σημαντικό να μην υπάρχει αποκάλυψη των απορρίτων, των επιχειρηματικών απορρίτων. Εδώ λοιπόν μπορώ να δείξω ευελιξία, αλλά δεν είναι δυνατόν στην τελική ανάλυση αυτή η πρόταση να επιδεινώσει ακόμα την κατάσταση περαιτέρω για τους παραγωγούς γενώσιμων. Προσβλέπω στη συζήτηση και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να δούμε τι θα πούν και οι άλλες δύο Επιτροπέ που γνωμοδοτούν, αυτό ενδεχομένω να επηρεάσει και τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ. Και ξέρω ότι οι συνάδελφοι θέλουν να ξεκινήσουμε τι ψηφοφορίε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να πω δύο λόγια, γιατί δυστυχώ θα χάσω την, ε, συζήτηση, την συνάντηση των σκηνοδών την Τετάρτη. Δεν είναι μυστικό ότι οι πράσινοι, ότι η ομάδα έχει σημαντικές αμφιβολίες για την ε, χρησιμότητα του συστήματος SPC, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να παρατείνει τεχνητά την προστασία για επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τα διπλώματα βρυστεχνίων, ακόμα και για εταιρείες που δεν έχουν επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη των ε, φαρμάκων αυτών. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί. Συμφωνούμε ότι αυτή η πρόταση δεν θα μπορέσει να λύσει όλα τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα είναι ένα μικρό βήμα, αν θέλετε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά εντός των όσων προσπαθεί να πετύχει αυτή η πρόταση, θεωρώ ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα θέματα πρόσβασης στην αγορά για τα γενώσιμα φάρμακα και αυτό περιλαμβάνει το stockpiling, τη φύλαξη σε ό,τι αφορά την δυνατότητα εφαρμογή της απαλλαγής από το SPC και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. σω δεν είναι το σωστό σημείο να επισέλθουμε σε λεπτομέρειε. Μπορούμε να το βάλουμε σε μια ρήτρα αναθεώρηση σε ό,τι αφορά το σύστημα SPC, ότι θα πρέπει να εξεταστεί πιο εντελεχώ στο μέλλον. Αυτό φυσικά δεν ε, πρέπει να εμποδίσει την ολοκλήρωση τη πρόταση αυτή στην τρέχουσα θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Όπως ε, είπα και πριν, χαιρόμαστε για το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Πιστεύουμε ότι είναι αρκετά ισορροπημένο, έχει αρκετές ισορροπημένες ιδέες. Όσον αφορά τις επιπλέον τροπολογίες, κατά τη γνώμη μας υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό, για παράδειγμα όσον αφορά την κοινοποίηση όπου για μας δύο στοιχεία είναι κλειδί. Αφενός πιστεύουμε ότι όποιος έχει συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας πρέπει να ενημερώνεται όσο χρειάζεται για να μπορέσει να ελέγξει κατά πόσο υπάρχει παραβίαση ή όχι του συμπληρωματικού του πιστοποιητικού προστασίας. Αυτό αφενός. Αφετέρου όμως πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει ε, μεταφορά ευαίσθητων εμπορικά πληροφοριών. Και αυτή την οπτική γωνία πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια της πρότασης αυτής. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς προτιμήσαμε την πρόταση της δημοσίευσης που είναι προς το συμφέρον όλων. Η διαφάνεια και αντικειμενικότητα είναι καλύτερη εγγύηση για παραπλάνηση κτλ να μην υπάρχει παραπλάνηση κτλ. Τώρα, ε, πιστεύω ότι θα μπορέσει να υπάρξει ένας συμβιβασμός που να περιλαμβάνει τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Εκεί που διαφωνώ όμως είναι ότι όταν ακούω πως δεν είναι προς το συμφέρον των ασθενών η πρόταση αυτή. Μα πρόκειται για παρέκκληση για τις εξαγωγές, αλλά δεν πρόκειται για ασθενείς τρίτων χωρών. Πρόκειται για να διασφαλίσουμε ότι δημιουργούμε αρκετές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας της Ευρώπης, γιατί θέλουμε ακριβώς οι επιχειρήσεις αυτές να παραμείνουν στην Ευρώπη και να έχουν μια πολύ καλή θέση στην Ευρώπη. Να επιβεβαιωθεί η θέση της Ευρώπης δηλαδή ως κόμβος για τις ε, φαρμακοβιομηχανίες. Συνεπώς πρέπει και η έκθεση αυτή να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς να φροντίσουμε οι επιχειρήσεις μας να μην φεύγουν, να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό ε, για να προχωρήσουν με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αν μια επιχείρηση μείνει στην Ευρώπη και ξεκινήσει και την παραγωγή στην Ευρώπη, θα είναι έτοιμη όταν χρειάζεται και θα έχει και την ευκαιρία να προωθήσει τα προϊόντα της στην Ευρώπη. Δηλαδή ενισχύεται η θέση της απέναντι σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Συνεπώς, θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για μια πρόταση που συνεισφέρει στην πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα. Υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρησης. Προτείναμε να δούμε τι βελτίωση θα έχει προκύψει. Και έτσι πιστεύουμε ότι η εξαίρεση αυτή για τις εξαγωγές μπορεί να πετύχει τους στόχους της πρότασης με ισορροπημένο τρόπο, χωρίς να κινδυνεύουμε, κάτι το οποίο θέλαμε να αποφύγουμε με τις ρήτρε ασφάλειας, να υπάρξει στρέβλωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ωραία, συνεπώ μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και συνεχίζουμε και περνάμε στις ψηφοφορίες. Έχετε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας σας φαντάζομαι μαζί σας. Σωστά. Αρχίζουμε λοιπόν με το σχέδιο έκθεσης υπομορφή επιστολής για την ψηφιακή αγορά. Ο κύριος Φω είναι ο εισήγητη. Άξελ πρόκειται για μια νέα μοναδική ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Φω. Σχέδιο γνωμοδότησης τώρα, ασφάλιση καταστικής ευθύνης όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα. Τροπολογία αριθμό 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για τη 18 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 23. Ψηφίστε. Απορρίφθηκε. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε 27. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά.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 ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σχέδιο γνωμοδότησης τώρα, τροποποιημένο, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια, κυρία Μπερζερό. Συνεχίζουμε τώρα με τη δικιά μου έκθεση που έχει να κάνει με τους ε, ισχυρισμούς για διασυνοριακές ε, επιστροφές έργων τέχνης κλπ. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτη. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, 25 γνώμη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Εγκρίθηκε νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Εγκρίθηκε. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε την 33 παρακαλώ. Απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 και κουλ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε τη 42 παρακαλώ. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε τη 44. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Τη 49 μάλλον απορρίπτεται. 48 διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 55 απορρίπτεται Κούλτη 12 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Τα. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται κουλτ 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται όχι, είναι Στο Κουλθ 4 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Καταπίπτει. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτή καταπίπτει. 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 και κουλτέντεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτη 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 85 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε την 85, εγκρίνεται, 86 έχει αποσυρθεί. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κούλτ 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 93. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κάλτε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 και κουλτένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει επομένως ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης το σύνολό σύνολο της συγγνώμη. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και <laughs> αυτή ήταν άλλη μια ευκαιρία να συγχαρώ τον εαυτό μου. Στο τέλος τώρα πάμε στην απαλλαγή της εφαρμογής του Γενικού Προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 8 ελέγχουμε παρακαλώ Μάλιστα, δεν είχα δει. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορείς να ελέγξουμε και την 9, παρακαλώ. Μπερδεύτηκα. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πολύ ωραία. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 14. Εγκρίθηκε. Και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Πολύ ωραία. Thank you. Uh, we continue... Σας ευχαριστώ και συνεχίζουμε με την έκθεση του κ. Κοφεράτη για την επίδοση εγγράφων. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 και 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 65. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Μία ψήφος λείπει. Εγκρίθηκε. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ και 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Ω, συγγνώμη. Και πάλι. 112 την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη ε, η 35 απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος 113 υπέρ καταπίπτει 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Okay. My, my Να επαληθεύσουμε την 36 παρακαλώ. Γιατί υπήρξε έτοιμα για ηλεκτρονικό έλεγχο. Για την 36 παρακαλώ. Ελέγχουμε την 36. Απορρίφθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε και την προηγούμενη. Πρέπει να την ψηφίσουμε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 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 και 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Καταπίπτει. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το σχέδιο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά παρακαλώ τώρα. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κομφεράτη. Συνεχίζουμε. Σχέδιο έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή υποδείξεων σε αστικέ και εμπορικές υποθέσει Ράντεφ, συμβαστική 1, υπέρ, κατά, απόχέ, έγκρινεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 49, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Η 50, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51, υπέρ, κατά, Απόχε εγκρίνεται. 53, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ καταπίπτει 54 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ ελέγχουμε το 54 τέλεχος για το 54 παρακαλώ απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά. Να αλλάξουμε παρακαλώ την 14. Εγκρίθηκε. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την 73 εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 1 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 25 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η έκθεση στο σύνολό της ηλεκτρονικά εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Στον κύριο Ραντεφ, ο οποίος είναι απόν, βέβαια. Και τώρα έχουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης για μια βιομηχανική πολιτική σε ό,τι αφορά την ε, ρομποτική και την ραμπινεμοσύνη. Ε, Μία μόνο ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια στην κυρία Ντελβού. Τώρα περνάμε στην έκθεση αναθεώρησης στις αναθεώρησης στα ρίκα μάλλον και πάλι ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκαν. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκέριγκερ. Μήπως έχουμε τίποτα άλλο. Επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 23 Ιανουαρίου. Μα, συγγνώμη, είναι η πιο σημαντική ανακοίνωση, λέει ο πρόεδρος. Να σας καλέσω. Στο δείπνο της Επιτροπής ε, Λόου C2 c αύριο στις 7 αύριο κατά πάσα πιθανότητα τότε θα σας πω χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα Be the case. I wish it now. Thank you. Αν δεν καταφέρετε να έρθετε, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα τώρα.